γίνεται δεκτή. Δεν ξέρω τώρα, με συγχωρείτε, εσείς τι θέλετε. Λάθος, παρεξήγηση. Λοιπόν, γκρίνεται αυτή η παράταση της Επιτροπής και προχωράμε στην έκθεση για την θνησιμότητα ε, λόγω αλίας, ε, ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Επόμενο. Η έκθεση Γκέριγκερ. Και εδώ ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεκτή. Τώρα, ε, της κυρίας Μπενγκίν έχουμε δύο. Ψηφίζουμε τώρα για την Ελβετία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ευρωπαϊκή Ένωση Ελβετία. Έκλεισε ψηφοφορία. Δεκτή. Επόμενη επίση έκθεση τη κυρία Μπενγκίν Ε, πρόκειται για τη συμφωνία με την Νορβηγία. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Έκθεση Βέγγα σε ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Επόμενο. Έκθεση Αγγιλέρα Γκαρσία. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Επίσης δεκτή. Επόμενη έκθεση του κυρίου Καπούτο, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Επίσης εγκρίνεται και η έκθεση αυτή. Ε, έκθεση Ρόνταστ το πολιετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας. Εδώ υπάρχει πρόταση να απορρίψουμε την πρόταση Επιτροπής. Ψηφίζουμε γι' αυτό με ανατασχυρός υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ή απορρίφθηκε. Και δίνω τώρα, μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος, λάθος έκανα, προχωράμε, ονομαστική ψηφορία, Ζητώ συγγνώμη, πάλι λάθος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Χάζενκάμπ και ζητώ και συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επικαλιστώ το 9-3 θα ψηφίσουμε για τις ε, τροπολογίες για την Ολομέλεια. Πριν ψηφίσουμε για τη συμβαστική πρόταση, η δική μου η πολιτική ομάδα ε, θέλει να γίνει ψηφορία. Αυτό το σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα επιτρέπει την υπεραλίευση και αυτό αντιβαίνει στους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν έχει και καμία σχέση με την εντολή που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, οι διεθνείς οργανισμοί ζητούν να καταψηφιστεί το σχέδιο αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ βοηθήστε Βοηθήστε την αλία, βοηθήστε την διακήρυξη των ποικιλιών στη Βόρεια Θάλασσα κατά τη υπεραλήψη. Υπέρ. Υπέρ. Μισό λεπτό, ξανά λέω ο Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Μάλλον έκλεισε η ψηφοφορία. Έγινε δεκτή η πρόταση αυτή. Sorry, I ε, ε, λέει ο πρόεδρο. Λοιπόν, να σα εξηγήσω. Ψηφίσαμε για την ε, πρόταση της κυρία Χάζενκαμπ. Ξαναψηφίζουμε για την πρόταση τη κυρίας Χάζενκαμπ. Υπέρ, παρακαλώ. Υπέρ, λέει ο πρόεδρο. Είναι ονομαστική η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τώρα συνεχίζουμε με ονομαστική ψηφορία για το 183 ψηφίζουμε. 103 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Ξανά. Ξαναψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Έκλεισε η ψηφοφορία. δεκτή. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 1.04 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και τώρα πάμε στην έκθεση Μωράν Σαρτιέ και ε, Γιονγκέριους. Ο κύριος Μαρτά ζήτησε το λόγο και τον έχει κιόλας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αμφισβητώντα ε, τα όσα μάθαμε από τον τριμερή διάλογο και όσα προέκυψαν από εκεί, θέλουμε να ψηφιστούν όλες οι τροπολογίες. Παρακαλώ. Λοιπόν, να ψηφίσουμε διανάτες ισχυρό, υπέρ, κατά, αποχέ απορρίφθηκε. Άρα προχωράμε με ονομαστική ψηφοφορία για την 139. Ψηφίζουμε παρακαλώ. 39. Ε, ε, Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή και τώρα θα ψηφίσουμε διανατάσεως της χειρός για την 54. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. We now proceed with the vote Ψηφίζουμε τώρα για την έκθεση Engstrom. Είναι ε, ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η επόμενη. Έκθεση Scott Cato. Και πάλι ονομαστική ψηφορία. Με ονομαστική ε, ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, πριν από λίγο μας δόθηκαν κάποια πολύ περίπλοκα θέματα. Οι περισσότεροι βουλευτές δεν κατάλαβαν τίποτα και όταν ψηφίσαμε για την απόσπαση των εργαζομένων δεν είχαμε καταλάβει τι ψηφίζουμε. Εσείς είπατε ψηφίζουμε αλλά δεν είπατε τι ψηφίζουμε. Σας παρακαλώ να λέτε τι ψηφίζουμε, για ποιο πράγμα ψηφίζουμε και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υπάρχει σαφήνεια. Ε, δεν είναι έτσι, λέει ο πρόεδρος, δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Εγώ είπα για ποια έκθεση ψηφίζουμε, νομίζω ήμουν απόλυτα σαφής, ψηφίσαμε και ε, προέκυψε και πλειοψηφία και προχωράμε τώρα με την ψηφοφορία για την έκθεση Γκούτελαντ, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. The vote is ψηφοφορία. Δεκτή. Τελειώσαμε με τις ψηφορίες, προχωράμε στις αιτιολογήσεις ψήφου ε, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω όσοι επιθυμείτε να εγκαταλείψετε την αίθουσα ησύχως. Κύριε Κοέλιο, ε, διαδικαστικό. Κυρία Τόγια. Συνάδελφοι, εάν δεν συμμετάσχετε στην επεξήγηση ψηφών, παρακαλώ να φύγετε από το ημικύκλιο. Ε, κυρία Τόγια, πρόεδρε, για τη διαδικασία, ε, στην αρχή της Συνόδου Ακούσαμε, μια, ε, ακούσαμε λόγια που πραγματικά μας σοκάρισαν για ε, την κατάσταση που επικρατεί πολιτικός σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έπρεπε να είναι σεβαστή. Δεν μπορεί να εκφράζονται τέτοια λόγια που δεν αρμόζουν στην Ολομέλεια. Ήταν πολύ σοβαρά αυτά που υπόθηκαν. Θέλω να επαναλάβω εδώ, Πρόεδρο, ότι η χώρα μου είναι χώρα με το δικό της σύνταγμα, με πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ε, εγγυήθηκε το σεβασμό του συντάγματος κατά των επιθέσεων όσων θέλαν να αποδιγετήσουν το Σύνταγμα αυτό Είμαστε, και να το ποδοπατήσουν. Είμαστε ένα κράτος δικαίου. Ε, η Ιταλία αυτή τη στιγμή αυτό απέδειξε. Η πολιτική ε, διελκυστήντα από το είδου είναι απαράδεκτη. Στο Κοινοβούλιο να ακουστεί και πάλι ότι είμαστε κράτο δικαίου. Δεν μπορείτε να γίνεται επίθεση κατά των δημοκρατικών θεσμών με τέτοιο άνανδρο τρόπο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε, το καταγράφουμε, αλλά Όπω είδατε αφαίρεσα το λόγο από τον συνάδελφο, δεν ήταν διαδικαστικό, έκλεισα το μικρόφωνο του συναδέλφου, τον διέκοψα, οπότε ε, το θέμα αυτό μπορούμε να το δούμε περαιτέρω, αλλά το μικρόφωνο κόπε και δεν υπήρχε διερμηνία και δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τη συνέχεια στα Ιταλικά. Ε, ε πάντως την παρατήρησή σα την καταγράφω και θα ληφθεί υπόψη. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε το λόγο από τον συνάδελφο. Και περνάμε τώρα στην επεξήγηση ψήφων. Πρώτη, έκθεση Αγγιλέρα Γκαρσία. Για δύο λεπτά η κυρία Νταμάτο. Παρακαλώ.